προφανώς εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία. Κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, ε, ε, θα έχουμε εξηγήσει ψήφων όσον αφορά την, όσον αφορά την Επιτροπή αλίας. Έχει αλλάξει ο κανονισμός της αλίας όσον αφορά τη βιώσιμη αλία στην ε, Μεσόγειο. Η προθεσμία θα αρχίσει να ισχύει από αύριο. Τα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο ε, και μάλιστα στην αρχή της προσεχούς συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα διαβιβάσουμε όλα τα ψηφίσματα όσα έχουν εγκριθεί στα όργανα τα οποία αναφέρονται στα εν λόγω ψηφίσματα. Ε, λύεται η σημερινή συνεδρία.